το τέλος της ΣΟΑ ο αντισημιτισμός αυξάνεται και πάλι στην Ευρώπη. Ο ορισμός του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για την ανάμνηση του ολοκαυτώματος που εγκρίναμε το 2017 πρέπει να καλύπτει και καλύπτει τα πάντα. Επίσης δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις στα άτομα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή των χαρακτηριστικών φύλου και να τους αρνείται η, αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι στο κέντρο της πολιτικής μας, διότι ο ανθρωπισμός μιας κοινωνίας μετριέται από το πώς αντιμετωπίζει τις μειονότητες που περιέχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέλγα Στίβενς. Πρόεδρε, συνάδελφοι, Άκουσα τις ε, επικρίσεις για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, τα άτομα ΛΟΑΔ και οι γυναίκες. Δεν θα υπερψηφίσουμε την έκθεση παρά το ότι είναι σημαντικά θέματα. Αλλά είμαστε υπέρ και μια βοήθειας για τα άτομα με αναπηρίες. Η έκθεση όμως αυτή δεν κάνει σωστά τις διακρίσεις μεταξύ της ε, παράνομης και της νόμης μετανάστευσης. Η οικογενειακή επανένωση θεωρείται μέτρο, είναι μέτρο που ευνοεί την μετανάστευση. Και ε, μιλάμε υπερβολικά για τις πολιτικές ε, ασύλου. Όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια αυστηρή πολιτική για την ε, μετανάστευση. Είναι ένα συνονθήλευμα αυτή η έκθεση. Εγώ θα προτιμούσα τα θέματα αυτά, όπως πάντα προτείνουμε, να αντιμετωπίζονται χωριστά. Επίσης στην έκθεση δεν βλέπω να αναφερόμεθα ε, στο σκάνδαλο των πολιτικών κρατουμένων στην Ισπανία. Πώς είναι δυνατόν. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Η κυρία Ναταλή Γκρισμπέκ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2017 ήταν ε, ζωφερό έτος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδιαίτερα για την ελευθερία έκφρασης. Πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά, στο σώμα μας Χρειάστηκε να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή για να ε, τιμήσουμε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ασκώντας το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Αυτοί οι πρωταγωνιστές δημοκρατίας ε, που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου δολοφονήθηκαν γιατί έδειξαν πολύ κοντά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, το ξέπλυμα χρήματος και την φοροαποφυγή. Θα ξεχάγουμε τα συμπεράσματα που θα έπρεπε για την ελεύθερη έκφραση. Ενώ τώρα που ακούμε ανησυχητικές ρητορικέ κατά των μέσων ε, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπου υπάρχει, υπάρχουν επιθέσεις και εκφοβισμοί των υπερασπιστών των δικαιωμάτων. Πρέπει να θυμηθούμε τον Μπομαρσέ που έλεγε χωρίς την ε, ελευθερία να επικρίνουμε δεν μπορεί κανείς και να επενέσει. Στηρίζω την έκφραση, την έκθεση αυτή που καταδικάζει τις ε, υπερβολικές παραβιάσεις ε, του 2017 αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ράιντκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξουμε γύρω μας. Παντού στην Ευρώπη κατεβαίνουν στο δρόμο οι πολίτες, ε, είτε είναι Βουκαρέστη, Βουκουρέστη, είτε είναι Βαρσοβία, είτε είναι Βιέννη, είτε Βαρολίνο, κουνώντας οι μέσες της Ένωσης, απευθυνόμενοι σε εμά. Γιατί το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα Υφίστανται επιθέσει σε πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να υπάρξει δράση από την πλευρά μας. Το άρθρο 7 ε, απεδείχθη ισχυρό όργανο, αλλά παράλληλα στην εφαρμογή του είναι δύσχριστο συχνά. Και γι' αυτό θέλουμε επιπλέον δυνατότητες, εργαλεία για να στηρίξουμε το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των συμπολιτών μας. Για παράδειγμα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που να παρακολουθεί συνεχώς ε, την εξέλιξη του κράτους δικαίου. Να το συζητάμε συχνά το θέμα αυτό. Και αν υπάρχουν παραβιάσεις, να υπάρχει ένας μηχανισμός κυρώσεων για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο απευθείας εκλεγμένο όργανο των Ευρωπαίων πολιτών. Στην καταπολέμηση των ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να παίζει τον κύριο ρόλο. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με κάποια κράτη ή με κάποιες πολιτικές ομάδες. Είναι θεμελιώδης προσπάθεια όλων μας. Ας το κάνουμε λοιπόν από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δεχθείτε μία μπλε κάρτα από την κυρία Γραπίνη. Και μην καθυστερείτε γιατί έχουμε ψηφοφορίες σε λίγη ώρα. Μάλλον ναι, δεν μπορούμε να δεχθούμε τις μπλε κάρτες. Δίνω το λόγο στον κύριο Έθεριτζ. Μάρουσικ, δεν είναι εδώ και ο Στέθεριτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως και τα φυσικά δικαιώματα, περιλαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Να υπογραμμίσω μια λεπτομέρεια σχετικά με την ιδιοκτησία. Αυτό το οποίο κερδίζεις είναι η ιδιοκτησία σου. Υπάρχει το φυσικό δικαίωμα το να διαθέτει κανείς ελεύθερα τον καρπό της προσπάθειάς του. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της ιδιοκτησίας, το έσοδο αυτό παραβιάζεται μερικές φορές από τους εργοδότες. Είναι κοινή ε, πρακτική δυστυχώς να κατάσχονται οι ιδιοκτησίες για φορολογικά χρέη, αλλά είναι ανήθικο κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς όμως ε, έτσι συμβαίνει. Τιμωρείται ο κόσμος γιατί κάνει το καλό. Ο κόσμος επίσης πληρώνεται μερικές φορές και ανταμείβεται όταν κάνει κάτι το άχρηστο. Αυτό είναι πάρα πολύ άχρηστο πράγματι και εις βάρος της παραγωγικότητας της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν θα εξαφανιστεί, γιατί τι είναι η Ευρώπη, είναι ένα παράσιτο, αλλά το πραγματικό σώμα πάνω στο οποίο ζει και το απομιζά δεν πηγαίνει καλά. Κύριος Φουντούλης. Εδαφικότητες που αναφέρει περιέχει και μία πρόταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Σας τη διαβάζω αυτολεξή. Πρόληψη κάθε διάβρωση του κράτους δικαίου, το οποίο δεν είναι η άνεφορον εφαρμογή των νόμων, αλλά η δημοκρατική αποδοχή της υπαγωγής σε νόμους αντιθέτω το θεμέλιο του κράτου δικαίου είναι ακριβώ η ανεφόρον εφαρμογή των νόμων. ποιο ορίζει του όρου υπό του οποίου θα εφαρμόζονται οι νόμοι; ελπίζω ο συντάκτη εκθέσεως να μην θεωρεί πω τα ευρωπαϊκά όργανα ή οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν τέτοια εξουσία. επιπλέον πολλή λόγο γίνεται για τα δικαιώματα των λαθρομεταναστών και των μειονοτήτων. αρχικά α ξεκαθαρίσουμε πω η μετανάστευση δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. αντιθέτω τα κράτη έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν οποιοδήποτε μπορεί να περάσει τα σύνορά του ακόμη σχετικά με τι μειονότητε είμαι αντίθετο σε οποιαδήποτε πρακτική θετικών διακρίσεων. τα μέλη μειονοτήτων πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσει όπω και οι υπόλοιποι πολίτε των κρατών τίποτα παραπάνω. τέλο να σα θυμίσω πω ποτέ αυτό το σώμα δεν καταδίκασε έστω και μία από τι εκατοντάδε επιθέσει εναντίον εθνικιστών. ω πατέρα ενό παιδιού δολοφονημένου από τρομοκράτε τη αριστερά δικαιούμαι να σα ονομάζω υποκριτέ. Ευχαριστώ. Επόμενος ο μιλητής ο κύριος Βέρα. Θέλω να συγχαρώ... Όχι, δεν θα μπορούσα να είμαι σύμφωνος γιατί εδώ υπάρχει μια διάβρωση της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξαιρούμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και η παράνομη μετανάστευση γίνεται αρετή και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τόπος όπου όλοι φύστανται βία, οι γυναίκες, οι πάντες. Αυτό δεν ισχύει. Είμαστε χώρος ελευθερίας, ισότητας με το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στον κόσμο. Που όλοι το εκτιμούν. Γιατί κατά τη σύνταξη αυτή τη έκθεση δεν συζητήσατε περισσότερο με του συναδέλφου, Γιατί δεν επιδιώξατε ευρύτερου συμβιβασμού, γιατί ε, χρειάστηκε να γίνουν ε, κατά την παράθεση ψηφοφορίες. Δεν νομίζω ότι είναι συμμετρική, ισορροπημένη αυτή η έκθεση, δεν είναι αντικειμενική και δεν θα τη στηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάιντενχολτσα. Ευχαριστώ πολύ. Η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ετήσιας δραστηριότητας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν ε, τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και πώς είναι η κατάσταση στα, συγκεκριμένα, στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και πώς ε, εξελίσσεται η κατάσταση. Ο εισηγητής Τερικάπρας ε, έθεσε ως καθήκον να ασχοληθεί συστηματικά με αυτό το θέμα και το επέτυχε αναμφίβολα και τον συγχαίρω. Σωστά τονίζει το ρόλο της, ε, του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η εμπειρογνωμοσύνη της πρέπει να αξιοποιείται περισσότερο και για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης, αλλά και ως σώμα εμπειρογνωμόνων κατά την εκπόνηση νομοθετημάτων. Η ομάδα μας συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις. Θα ήταν πολύ σκόπιμο ο οργανισμός αυτός και με δική του πρωτοβουλία να μπορεί να δράσει. Θα έπρεπε όμως για να γίνει αυτό να υπάρχει επαρκές προσωπικό και ε, προϋπολογισμός. Η Μπόνικα Μακοβέη. Να πάρω. Mm. στο Αζερβαϊτζάν οι δημοσιογράφοι κινδυνεύουν τη ζωή τους και την ελευθερία τους για να γράψουν και να εκφραστούν ελεύθερα. Χουσεϊνόφ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για συκοφάντηση τον Μάρτιο του 2017 αφού δημοσίευσε ε, διάφορα είδη πολυτελείας που ανήκανε σε βουλευτές. Κάνει απεργία είναι με άλλους πολιτικούς ε, φυλακισμένους και ε, ανθρώπους που υπερασπίζονται τη συνείδησή τους. Ε, Βεβαίω έχουν επινοηθεί οι διάφορες παραβιάσεις και έχει αρχίσει μια έρευνα ε, και τώρα έχει μεταφερθεί, έχει συλληφθεί ε, και κάνει ακόμα απεργία πείνας σήμερα. Γι' αυτό κάνω έκκληση στην κυρία Μογκερίνη ούτω ώστε να έχει μια αντίδραση καθαρή όπως είχε αντιδράσει κατά την πρώτη σύλληψή του. Η ζωή και η ελευθερία δεν είναι διαπραγματεύσιμα, γι' αυτό ζητάω ε, σύντομα να ελευθερωθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Σοζίτενβελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι ορισμένες παρεμβάσεις δείχνουν ε, σαφώς πόσα περισσότερα πρέπει να επενδύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα αξιών. Και ακούω ε, τους συναδέλφους που λένε «Μα γιατί δεν έχετε περισσότερους συμβιβασμούς, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συμβιβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για μερικές βασικές αρχές» λέτε «Α, όλα είναι πάρα πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει διακρίσεις κατά των γυναικών». Πόσες γυναίκες στην καθημερινή του ζωή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν βία και αυτό δείχνει πόσο χρειάζεται ε, να υπερσπιστούμε τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ. Ε, έχουμε στην χώρα μου 200 ε, υπουργού ε, που 200 χριστιανούς οι οποίοι έχουν δηλώσεις ομοφοβικές. Ε, ποιος άλλος έχει υπογράψει τέτοιες δηλώσεις όπως αυτή η Θα ήθελα στην ε, στην αιτιολογική σκέψη 7 και παράγραφο 23 να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα των γυναικών να αποφασίζουν για την δική τους την μοίρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση αρχών και αξιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτη και ανυποχώρητη στην εφαρμογή των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο για τι χώρε μέλη τη, αλλά και για τι χώρε που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μα είναι απαράδεκτο και αδιανόητο χώρε που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίε λαμβάνουν και προενταξιακή βοήθεια, δηλαδή επιβραβεύονται κάθε χρόνο, όπως είναι η τουρκία να παραβιάζουν συλλήφθη το κράτος δικαίου τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης τους διεθνείς νόμους και συμβάσεις να παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και να επιβραβεύονται μέσα από την ευρωπαϊκή ένωση προσφέροντας τους χρηματοδότηση προγράμματα προενταξιακή βοήθεια. εάν ερωτηθούν οι ευρωπαίοι πολίτες εάν σε χώρες όπως η τουρκία αλλά και η Αρβανία που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο εάν θέλουν να χρηματοδοτούν αυτές τις χώρες που παραβιάζουν αρχές και αξίες η απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών θα είναι όχι. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το μήνυμα ότι είναι ασυμβίβαστη σε αυτά και πρέπει να επιβληθούν μέτρα και κυρώσεις για να γίνουν αντιληπτά όλα αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφανο Μάουλου. με λάθος τρόπο αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεται κυρίως στον τομέα της μετανάστευσης με δύο αρχές οι οποίες τροφοδοτούν και δημιουργούν συνθήκες παρανομίας. Λέει ότι η μία πόθηση είναι μία λύση. Οπότε θα πρέπει να υποδεχθούμε όλους όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και το κάνει αυτό με ακόμα χειρότερο τρόπο όταν λέει ότι οι ΜΚΟ πρέπει να υποστηριχθούν. Αυτό είναι αντίθετο με την πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει στη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα, θα έλεγα, πλοκάμι παρανομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και δυστυχώς τροφοδοτείται αυτό το πλοκάμι παρανομίας από την Αφρική και Δίνουμε εκατομμύρια βέβαια στην Βόρειο Αφρική, σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα και γι' αυτό θα καταψηφίσω την έκθεση που δεν είναι διόλου πραγματιστική. Ευχαριστώ η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Εντάξει. όπως λέει η έκθεση, Πρέπει να βασιστούμε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, την, τον διαχωρισμό των εξουσιών και το κράτος δικαίου. Όμως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και συμφωνώ ότι το άρθρο 7 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν αποτύχουν όλες οι άλλες προσπάθειες. Θα πρέπει να είναι ίστατη καταφυγή. Όμως ε, υπάρχουν κάποια θέματα με τα οποία δεν συμφωνώ σε αυτή την έκθεση. Για παράδειγμα ότι πρέπει να γίνεται αυτή η μονομερής αποτίμηση των ΜΚΟ στη Μεσόγειο. Ορισμένα που λέγονται είναι σωστά. Αλλά είναι δυνατόν έτσι να ευνοούμε την παρόν μετανάστευση και τους διακινητές. Βεβαίω υπάρχουν ευάλωτα άτομα όπως οι μητέρε και τα μικρά παιδιά ε, στα ελληνικά νησιά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα για να βοηθήσει τα άτομα αυτά τον παρόντα χειμώνα. Είμαι κατά των ε, συστάσεων που υπάρχουν στην έκθεση για την επικύρωση τη συμφωνίας της ε, Κωνσταντινούπολη για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τη σεξουαλική υγεία. Η Ένωση θα πρέπει να προστατεύσει τη ζωή. Όχι το αντίθετο. Η κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο ε, περνάμε από τη διαδικασία έγκρισης αυτής της έκθεσης και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βασίζεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δίνουν και δεν προβλέπεται το δικαίωμα της ε, το δικαίωμα της έκτρωσης και γι' αυτό ε, εδώ θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε στην απόφαση της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης. Ε, υπάρχουν τέσσερις αναφορές στην έκθεση λοιπόν στο φύλλο, στον όρο φύλλο. Χρησιμοποιείται η λέξη φύλλο λοιπόν, χρησιμοποιείται επίσης επανειλημμένα η λέξη έκτρωση. Ε, στην ουσία αναφέρεται απλά στην ελευθερία συνείδησης και αυτό το οποίο προβλέπει ουσιαστικά η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ λοιπόν την πρόταση αυτή. Θα ξεκινήσω τη διαδικασία ε, Χώσε Φαρία πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Τερικάμπρα, στον οποίο συγχαίρω, αποδεικνύει ότι το 2017, 8 χρόνια μετά την έναρξη ισχύω τη ε, χάρτα, ε, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε βεβαίω ε, το πιο προχωρημένο στον κόσμο, αλλά η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η ομοφοβία, οι διακρίσει κατά των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίε, όλα αυτά εξακολουθούν να είναι σοβαρά προβλήματα. Σε μερικέ χώρε τη Ένωση, ε, διαπιστώσαμε σοβαρά προβλήματα διαφθοράς. Αλλά πώς μπορούμε να καταδικάσουμε ε, παραβιάσεις ε, σε τρίτες χώρες αν εμείς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για όσα συμβαίνουν στη δική μας επικράτεια. Πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες κυρώσεις για όλες αυτές τις παραβιάσεις. Αν το αγνοήσουμε δεν είμαστε σωστό κράτος δικαίου γιατί είμαστε εμεί οι κληρονόμοι του ανθρωπισμού και αυτό πρέπει να μας συνδέει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Τέρι Κάμπρας και τους κοιόδης εισηγητές για την προσπάθεια που έκαναν το 2017. Δυστυχώς δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στον τομέα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ισότητα των φύλων, η παραβίαση ε, των δικαιωμάτων των παιδιών, των ανηλίκων. Παραβιάζεται η αρχή ότι, ε, που λέγει ότι απαγορεύεται η κράτηση ανηλίκων ε, λόγω του ότι μπορεί να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προτάσεις οι οποίες γίνονται σε σχέση με τη βία για λόγους φύλου, για λόγους διάκρισης και εδώ υπάρχει σωστή παραπομπή στην απόφαση της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης. Ε, ε, μένει ο εισηγητής και στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το κράτος δικαίου και επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ Τόμασιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαβάζοντας την έκθεση αυτή μου διαμορφώνεται η αντίληψη ότι κάποιος που δεν είναι γυναίκα μετανάστης ή μειονοτικός δεν έχει δικαιώματα. Εμείς θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την αριστερίστικη ρητορική και να αναφερθούμε στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών. Υπάρχουν εκατομμύρια άστεγοι, υπάρχουν εκατομμύρια χρεωμένων, υπερχρεωμένων Ευρωπαίων Υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που ζουν μέσα σε μεγάλη φτώχεια και που οι γονείς τους δεν μπορούν να τα ταΐσουν σωστά. Η αξιοπρέπεια είναι λοιπόν το πρόβλημα του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο λείπει και εδώ και δυστυχώς πάρα πολλές φορές προωθούνται ε, τα δικαιώματα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς και με πολύ επιλεκτικό τρόπο όπως το δικαίωμα της μετανάστευσης. Ένα επιπλέον ομιλητή στα πλαίσια του ΚΑΤΣΤΙΑΙ και μετά θα περάσουμε στην παρέμβαση της Επιτροπής. Ο κύριο Επιτίδιος, ένα λεπτό. Ε, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται μεταξύ των άλλων αξιών ε, και, στην, ε, και στο σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων πολλά κράτη της παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά. θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού όμως σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνη η ευρωπαϊκή ένωση που συμβαίνει αυτή η κατάσταση διότι ε, αντιμετωπίζει με τρόπο επιλεκτικό τις παραβιάσεις αυτές. παραδείγματος χάρη ενώ έχετε κάποια κράτη να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ατιμωρητή τιμωρεί κάποια άλλα κράτη. ενώ κόπτεται και δικαίως για την ελευθερία τη δικαιοσύνης Εν τούτης, ανέχεται να φυλακίζονται για πολιτική σκοπιμότητα οι βουλευτές της Καταλωνίας και δεν αντέδρασε όταν στην Ελλάδα παραβιάστηκε αυτή η αρχή προκειμένου να διωχθούν ε, πολιτικά ο αρχηγός και οι βουλευτές του τρίτου σε δύναμη πολιτικού κόμματος της Ελλάδος της Αυγής. Υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου αλλά παράλληλα ποινικοποιεί την έκφραση της αντίθετης απόψεως χαρακτηρίζοντάς την ρατσιστική, ξενοφοβική και ομοφοβική πρέπει λοιπόν να απαλλαγεί από αυτή την ε, ε, υποκρισία η ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Χωρείτε, με συγχωρείτε, πρέπει να δια, διακόψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα κλείσουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Γιούροβα θα ήθελα να αντιδράσω σύντομα για τα όσα ακούσαμε, διότι απορρίπτω τα όσα λέχθηκαν για την επιλεκτική, και ε, τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Έπρεπε να αντιδράσω πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να συμπεράνω ε, από αυτήν την συζήτηση ότι πρέπει να αναφέρουμε το ρόλο της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε έχουμε τις ε, νέους κινδύνους ε, που αναπτύσσονται ε, και πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλήσαμε ε, πολύ για το χώρο ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, που έχει περιοριστεί για τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης που πρέπει να υποστηριχθεί. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένας χώρος για περαιτέρω συζήτηση για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Δεν μιλήσαμε για τη νέα τάση που είναι το μίσος και την προβληματική κατάσταση στο ίντερνετ. Ε, στα... Εκεί πρέπει να προστατεύσουμε τα άτομα που κινδυνεύουν. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω την συνέχιση της συζήτησης για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Σας παρακαλώ να, με ησυχία να λάβετε τις θέσεις σας και δίνω τώρα τον λόγο στον εισηγητή τον ε, Μαρία ε, Τερικάμπρα. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και την υποστήριξή σας. Με την έκθεση αυτή θα στείλουμε ένα μήνυμα ότι η πρόθεση και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας του κράτους δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να καταστήσουν την Ένωση μοναδική ε, στα, ε, στα πολιτικά της σχέδια μόνο θέτοντας την ευημερία των ατόμων στο επίκεντρο της πολιτικής και, και των αποφάσεων της Ένωσης θα μπορέσει η Ευρώπη να επανακτήσει σύνδεσμο με τους πολίτες της. Γι' αυτό ο χάρτης θέτει τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταγγέλουμε ε, τις παραβιάσεις των διαφόρων διατάξεων. Είναι ευθύνη μας να προστατεύσουμε τους πιο αδύνατους ε, και να αντιμετωπίσουμε το κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Έχουμε ξεπεράσει κατά ένα λεπτό και 49 δευτερόλεπτα το χρόνο μας και τώρα θα περάσουμε σε ένα λεπτό στην ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε. Θα ζητώ σε όσους είναι όρθιοι να καθίσουν, να εγκατασταθούν. Κυρίως ο κύριος Ανδριέ. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε καθίσει και αρχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Κουρουμπασέφ θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Ζήτησε το λόγο και του δίνω το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Κουρουμπασέφ. Δεν τον βλέπω να καταφθάνει. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Όχι, όχι, μην εκνευρίζεστε. Είναι με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε για την έκθεση αρκετή ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Μπέγκε. Έκθεση εφαρμογή σχετικά με τον εμπειρικό πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης με Κεντρική Αμερική. Μία μόνο ψηφοφορία, ον με ονομαστική ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα ψηφοφορία, Εγκρίθηκε. Περνάμε στην έκθεση των κυρίων Φερνάντες και Γκουαλτιέρη, θέσπιση του προγράμματος Invest EU. Αρχίζουμε με την τροπολογία 1 CP1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 1 CP2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένα CP3 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 1 CP4D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες Όχι, απορρίφθηκε, δεν εγκρίθηκε. Ένα CP5 σε δύο τμήματα. Πρώτος, υπέρ, πρώτο, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ένα CP6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ένα CP7 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι πολύ σαφή, σαφές το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 21D υπέρ, κατά, αποχές Απορρίφθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 1 CP8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Νομαστική ψηφοφορία για την 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 1CP9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 31, 31, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ένας CP10 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για τη 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 6 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Ένα CP11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για την 7CP1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε για την 1CP12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία. 7 CP2, 1 CP13, 15 CP2, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία 7 επί 3, 1 επί 14, 15 επί 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 7 επί 4, 1 επί 15, 15 επί 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 7 CP5, 1 CP16, 15 CP5, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορριφθήκε. Ψηφίζουμε για την 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 34 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 1 CP18 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. 35 με, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 22D υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 9D και 23D υπέρ κατά αποχές Ένα ένας CP19 ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 36 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορριφθήκε 10 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 37, πάντοτε ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε ονομαστικά για την τροπολογία 38 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία και τη 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε ονομαστικά για την 11, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 12, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για τη 13, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. απορρίφθηκε 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 2 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 1CP20. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 1CP21. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για τη 14. Αρχή η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε για την 1CP22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι πολύ σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 1CP22. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία για την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 18D υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 1 υπή 23, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 4D και 19D υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Ένας cp 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 20D, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 5 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε. Ονομαστική ψηφοφορία για την 5. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε λοιπόν για την ε, πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το 59-4 ζητώ το θέμα να παραπεμφθεί και πάλι ε, στην Επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε για αυτή την πρόταση. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίθηκε, παραπέμπεται και πάλι στην αρμόδια Επιτροπή το θέμα για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Γκάλ προσωρινό ταξιοδευτικό έγγραφο. Έχουμε τις τροπολογίες 1 ως 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 6. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά είναι περίπου το ίδιο θα ελέγξουμε για να μην υπάρξει λάθος για την 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχέσα νομίζω ότι εγκρίθηκε. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κουμπούλα Νάτρη πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ 2021-2025. Έχουμε την Επιτροπή στο συνολικά, το υπέρ κατά εγκρίθηκε. Πρώτο τμήμα, ε, τα πρώτες τροπολογίες υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε, με συγχωρείτε. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 602. Ποιος είναι πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο ε, τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ονομαστική ψηφοφορία για την 11 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε τροπολογία 16 ονομαστική ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίθηκε 34 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 5 Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5. πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε στην 31 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για την 32 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 33 με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε και κλείνουμε με την ε, ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε ε, στον έκθεση του κ. Μάτο, ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 3, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, ποιος ε, αποχές, Τέσσερα με ονομαστική ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Παράγραφος 10, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος 16, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, πάντα με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, ονομαστική ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική Πέρα της ψηφοφορίας. Κείμενο, δύο τμήματα, άρχεται ψηφοφορία ονομαστική πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία εγκρίθηκε δεύτερη ε, ονομαστική ψηφοφορία δύο τμήματα πρώτο τμήμα πέρα της ψηφοφορίας Απορρίφθηκε. Δεύτερο ε, τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ε, το παράγραφο C, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίθηκε ονομαστική ε, ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην εισήγηση του κυρίου Τόρβαλτσα, ε, Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση 2000. le Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση επί της τροπολογίας υπαριθμών 10. Τέλος. Η Γκουέ το έχει ζητήσει. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Δεν έχει ζητηθεί για την 12 ονομαστική κλίση. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, απερίφθη. Ονομαστική κλίση για το 13. Ψηφίζεται για την 13. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση για την 3. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση για το 4D. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απέχουν. Απερίφθη. 6 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη Επτά υπέρ κατά αποχές απερίφθη Οκτώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη ονομαστική κλίση για την τροπολογία 1 ψηφίζεται τέλος δεκτή τώρα για την 2 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά ποιοι απέχουν απερίφθη Ονομαστική κλίση για το σύνολο. Ψηφίζεται. Τέλος. Περνάμε τώρα σκέλα. Εμπορική συμφωνία Κολομβία και Περού. Τροπολογία 1. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Το 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 4. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαρίθμου 4. Τέλος. Δεκτή. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 18 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Ονομαστική κλίση για το δεύτερο τμήμα ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Για την πέντε ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση για την 6 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση για την τροπολογία 8 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση τώρα για το ψήφισμα στο σύνολό του. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Τελευταία έκθεση για την οποία έχουμε να ψηφίσουμε είναι η έκθεση Τερικάμπρας κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Λοιπόν, 7, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 10, ποιο είναι υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 7. Παράγραφος 7, δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτό. Αρχικό κείμενο παράγραφος 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αρχικό κείμενο παράγραφος 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ονομαστική ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 15. Πράγματι δεν είναι σίγουρο. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Δεκτή η παράγραφος 15. Λοιπόν, παράγραφος 23, αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Ψηφίζουμε για την 22, ονομαστική κλίση, ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Διολογική σκέψη F δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική κλίση. Μην αποσύρετε τις κάρτες σας ακόμα. Δεκτή. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι.